Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ας ξεκινήσουμε αμέσως, γιατί η ημερήσια διάταξη είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη. Και έχουμε και φιλοξενούμενους οι οποίοι έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν σήμερα το απόγευμα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια σε ό,τι αφορά το θέμα του διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα τη Επιτροπή και τη σύσταση τη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Καταρχήν, να καλωσορίσω την κυρία Γκρέσλε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τον κύριο Σβόμποτα από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια θα γίνει από κοινού, μια και οι τρει επιτροπέ μα έχουν μοιρασμένε αρμοδιότητε. Ιδιαίτερω καλωσορίζω την Έμιλι O'Reilly, Έμιλι την Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Παρακαλώ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η διερμηνία ε, δίδεται σε όλες τις ε, ε, γλώσσες εκτός από τσεχικά, φιλανδικά, ιστονικά, λιθουανικά και πορτογαλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες καλύπτονται. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ε, συνάντησης των συντονιστών θα σας ενημερώσω αργότερα ε, όταν ολοκληρωθεί η κοινή συνεδρία των Επιτροπών. Η Επιτροπή Αναφορών είναι η αρμόδια για τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και είναι χαρά μας Επανειλημμένως έχουμε φιλοξενήσει τον διαμεσολαβητή εδώ σε αυτήν την Επιτροπή για να συζητήσουμε τα απορίσματα και γενικότερα το έργο του, καθώς επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σήμερα θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις για την σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας ε, κατόπιν της έρευνας που έγινε σε ό,τι αφορά το διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής. Η σύσταση αυτή ε, δημοσιεύτηκε στις 31 Αυγούστου του 2018. Να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε ένα ψήφισμα για την ε, πολιτική ε, ακαιρεότητα της ε, Κομισιόν και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18 Απριλίου 18. Η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει το θέμα αυτό καθημερινά ανταποκρινόμενοι και σε αιτήματα και αναφορές πολιτών. Οι πολίτες ενδιαφέρονται γιατί ακριβώς έχουν προσφύγει στην Επιτροπή μας με αναφορές. Οπότε χαίρομαι που φιλοξενούμε στην Επιτροπή μας αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θα δώσω το λόγο καταρχήν στην κυρία Γκρέσλε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για τις εισαγωγικές της παρατηρήσεις και μετά στον κύριο Σβόμποντα από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Σεσίλια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ε, πρωτοβουλία που πήρατε για την ε, κοινή αυτή συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ε, θυμίσω αυτό που είχε ζητήσει κάποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διαδικασία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έχουμε δίπλωμα στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Λοιπόν, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια. Δεύτερον, ο εσωτερικό κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ακεραιότητα αντικειμενικότητα. Και τρίτον, η διαδικασία λήψη αποφάσεων στο Σώμα των Επιτρόπων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει αυτήν την ε, ακεραιότητα και αντικειμενικότητα. Αυτά είναι σημεία τα οποία απασχολούν και εμάς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχει διαμεραστεί στα ε, θεσμικά όργανα. Έχουμε Έχουμε ερωτήσεις για τις θέσεις ε, του Γενικού Διευθυντή και πώς αυτές θα πρέπει να επανδρώνονται και η μόνη θέση για την οποία δεν προκυρήσεται διαγωνισμό είναι η θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Για όλες τις υπόλοιπες υπάρχει ε, πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές ε, λοιπόν δεν γίνεται αυτό. Από το 2012 μέχρι το 2018 έγιναν 34 ε, εσωτερικές ε, μεταθέσεις σε σε ε, διοικητικές θέσεις εντός των θεσμικών οργάνων. Το άρθρο 4 του καταστατικού αναφέρει ότι πρέπει να κοινοποιείται κάθε διορισμός εγκαίρος και έχουμε ζητήσει να μειωθούν αυτές οι εσωτερικές μεταθέσεις στο ελαχιστό έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανοιχτού διαγωνισμού με υποψήφιους που θα πληρούν όλες ε, τις ε, προϋποθέσεις. Η, κυρία Γιάλα Σέντερ ε, θα είναι, είναι η, η συγγήτρια της σχετικής έκθεσης στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σβόμποντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει μετάφραση στα τσεχικά, έτσι. Είναι τα αγγλικά σας τόσο καλά, τόσο άψογα. Εγώ προσπάθησα να σε πείσω. Τώρα, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. και χαίρομαι που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτές μαζί με τις επιτροπές σας. Η επιτροπή στην οποία προεδρεύω είναι αρμόδια για τον κανονισμό προσωπικού και είχαμε συζητήσει τους, την τελευταία ε, είχαμε αποφανθεί επί της τελευταίας ε, τροποποίησης ε, του πλησιακού κανονισμού και άλλα συναφή θέματα. Δεν θα ήθελα να σπαταλήσουμε άλλο χρόνο. Όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να κάνουν περισσότερη προσπάθεια να εφαρμόσουν τις διατάξεις του υπηρεσιακού κανονισμού σε ό,τι αφορά τους διορισμούς σε Στι πιο υψηλέ θέσεις και γενικότερα σε οποιαδήποτε θέση, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες. Ευχαριστούμε και τους δύο συναδέλφους. Θα καλούσα τώρα την κυρία Ορέιλι να προχωρήσει με τη δική της παρουσίαση των πορισμάτων και των συστάσεων τους, δηλαδή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, μετά την ορισμό του νέου Γενικού Γραμματεία και θα δώσω το λόγο βεβαίως και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης τους συντονιστές ή τους αντικαταστάτες τους και αν έχουμε χρόνο μετά θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων με υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ, Έμιλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους πρόεδροι επιτροπών, αγαπητά μέλη, πολύ χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας εδώ σήμερα για να συζητήσουμε οποιαδήποτε ζητήματα ανακύπτουν από τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα. Χρειαζόμαστε διοίκηση που να συμμορφούνται προς τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Σε γενικές γραμμές η ενωσιακή διοίκηση πράγματι συμμορφούνται προς τα κριτήρια αυτά και τα υψηλά αυτά πρότυπα πολύ συχνά και γενικώ τα τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθεί συστάσεις από τον δικό μας ε, οργανισμό και από το Κοινοβούλιο σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν σε αυτούς τους διορισμούς. Είχαμε και τη βράβευση ε, πέρυσι ε, και περιμένουμε και νεότερες υποβολές και από το Κοινοβούλιο στα επόμενα χρόνια. Τώρα υπάρχουν κάποιες φορές κάποια προβλήματα και είναι ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα της ε, Επιτροπής να τα παρακολουθεί και γι' αυτό και δίδεται τόσο μεγάλη προσοχή σε αυτόν το θόκο. Εκφράστηκαν λοιπόν κάποιες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο του διορισμού. Ο διαμεσολαβητής άνοιξε μια έρευνα μετά από δύο καταγγελίες ε, δύο κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών του σώματο αυτού και περιμέναμε φυσικά το πόρισμα της δικής σας δουλειάς προτού ξεκινήσουμε τη δική σας ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ενδελεχή εξέταση χωρίς να υπάρχει καμία επικάλυψη. Μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον Απριλίο ξεκινήσαμε εμείς, εγώ, αποστέλλοντας γραπτές ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Ένα από τα ερωτήματα ήταν κατά πόσον η Κομισιόν είχε κάποια διδάγματα βγάλει από τις προηγούμενες εμπειρίες της. Η απάντηση ήταν ότι όχι. Αρνητική η απάντηση. Από εκεί πέρα προχωρήσαμε στην εξέταση των σχετικών εγγράφων. 8.500 σελίδες περίπου. Ήταν μια δύσκολη εξέταση και θα ευχαριστήσω και τις δύο συναρμόδιες υπηρεσίες για την τεράστια οργανωτική προσπάθεια. Θα πρέπει να πιέσουμε την Κομισιόν ώστε να εξετάσουμε όλο το σχετικό υλικό και να είμαστε σίγουροι ότι θα έχει καλυφθεί. Έχοντα πρόσβαση στα έγγραφα, ήταν σαφέ ότι πολύ λίγα από αυτά είχαν συνταχθεί πριν από τον διορισμό, με την τεράστια πλειοψηφία μετά τον διορισμό, ώστε να απαντήσουν διάφορα ερωτήματα του Κοινοβουλίου. Επομένω, από τον Αύγουστο, το τέλο Αυγούστου, είχαμε τα εξή πορίσματα. Πρώτον, ο κύριο Σέλμαϊερ είχε αρχικά συμμετάσχει σε μια δικασία πλήρωση σε ω Γενικού Διευθυντή. Όταν δημιουργήθηκε η κενή αυτή θέση, συμμετείχε και στην κοινοποίηση της καινής θέσης παρά το γεγονό ότι θα, μετά θα τον είχαν ενημερώσει σχετικά με την υποψηφιότητα αυτή τη θέση, κανονικά θα έπρεπε να έχει αποκλείσει τον εαυτό του από τι υποψηφιότητε αυτέ. Το γεγονό ότι δεν το έκανε δημιούργησε ένα κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων. Δεύτερον, όταν ο κ. Ζέλμαια υπέβαλε την υποψηφιότητά του, ε, απέκλεισε τον εαυτό του από την CCA, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για του Διορισμού, η οποία από εκεί και πέρα θα αξιολογούσε τους υποψηφίους. Αλλά προκειμένου να υπάρχει αναπληρωτής μεταξύ των ε, επικεφαλής διοικητικών δεν υπήρχε, ε, δεν είχε οριστεί, δεν υπήρχε χρόνος να οριστεί δηλαδή αναπληρωτής και επικεφαλής εξέτασης αυτής. Επίσης, η όλη διαδικασία 20 Φεβρουαρίου εκίνησε την ώρα του γεύματος αλλά η διαδικασία για τον διορισμό του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ολοκληρώθηκε μόνο αργότερα εκείνη την ίδια ημέρα, το οποίο δείχνει ότι η διαδικασία του διορισμού του Γενικού Γραμματέα δεν ακολούθησε το στόχο τη, ότι δηλαδή έπρεπε να πληρώσει μια γενή θέση, αλλά απλώ προσπαθούσε να εξασφαλίσει ότι ο κύριο Ζέλμαια θα ήταν επιλέξιμο προκειμένου να διοριστεί την επόμενη μέρα Γενικό Γραμματέα. Η Κομισιόν λοιπόν δεν χρησιμοποίησε τις ε, εξουσίες της αρμοδιότητες που έχει κατά ορθό τρόπο. Επίσης, με την έλλειψη της ενημέρωσης για την αποχώρηση του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα, ε, δημιουργήθηκε μια τεχνητή αίσθηση επίγοντος. Ιδιωτικά είχε ενημερώσει ότι θα αποχωρήσει μήνε πριν και θα μπορούσε να έχει ακολουθεί μια τελείως κανονική διαδικασία αναπλήρωσης. Επίση, ο πρόσωπος τύπου της Κομισιόν αντέδρασε με τρόπο λίγο ιδιότυπο, ε, έμεσο και συγκρουσιακό. Το οποίο βεβαίω είναι κατανοητό με όσα μάθαμε αργότερα σχετικά με το διορισμό. Ήταν αρκετά δύσκολο να λάβουμε ευθείε απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίζουμε αμέσω τα οποιαδήποτε και να έχουν ακολουθηθεί σε μια τέτοια σημασία διαδικασία και σχετικά με τα δικαιώματα του τύπου των μέσων ενημέρωση να έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με την όλη διαδικασία. Η σύστασή μα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να έχει διακριτή διαδικασία για το διορισμό του Γενικού Γραμματεία, διακριτή από άλλε αποπλήρωση άλλων κενών θέσεων, με ανακοίνωση και θέση εγκαίρω στην ημερήσια διάταξη του Κολεγίου των Επιτρόπων το οποίο θα πρέπει να διευρυνθεί για να συμπεριλαμβάνει και μέλη εκτό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μελλοντική πλήρωση θέσεων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κορυφαίε θέσει και η πλήρωσή του δεν θα γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών ή πολιτικών ομάδων ή κομμάτων. Και χαιρετίζουμε την πρόταση του Επιτρόπου Ότινγκα να υπάρξει μια διαθεσμική συζήτηση, διάλογο, που έλαβε χώρα 25 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι συζητήσει διαθεσμικέ δεν θα πρέπει να σταματούν την Κομισιόν από το να ακολουθούν τι συγκεκριμένε μου συστάσει σε σχέση με τον διορισμό, με την μελλοντική διαδικασία διορισμού του Γενικού Γραμματέα στο μέλλον. Περιμένουμε τι επίσημε απαντήσει τη Κομισιόν μέχρι 4 Δεκεμβρίου. Ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι η αξιολόγηση του κυρίου Ζέλμαια δεν ήταν αντικείμενο τη εξέτασή μα είναι ένας αξιωματούχος με άρτια προσόντα, έχει την εμπιστοσύνη του Προέδρου Γιούνκερ και αναλαμβάνει σε δύσκολους καιρούς η Κομισιόν ε, προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει επί τη βάση νομικών αιτιάσεων αλλά εμείς όπως και το Κοινοβούλιο υπογραμμίσαμε ότι ο διπλός διορισμός ε, μάλλον ξεπέρασε τα αρκετά ίδια ευέλικτα όρια που θέτει η νομοθεσία και οι διατάξεις για το διορισμό αυτό. Και δημιουργήθηκε ένα αρνητικό, μια αρνητική εντύπωση σχετικά με το πώ λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσει ύψη τη σημασία. Σε έναν κόσμο όπου ε, δημοκρατικέ ε, διαδικασίε και διατάξει απειλούνται, ε, η κοινή γνώμη στρέφεται προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τη συμπερασπίζεται. Δεν πρέπει λοιπόν να τροφοδοτούμε αφηγήματα που τελικώ είναι επιζήμια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ράιλι για το έργο σας και θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο επιτελείο σας γιατί ήταν τεράστιος ο όγκος των εγγράφων και η εξέτασή τους πρέπει να πήρε αρκετό καιρό. Τώρα θα ήθελα να καλέσω την κυρία Σούζαν Πάντερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο και να μας εκθέσει τις δικές της απόψεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίξτρομ. Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι εμιλητές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το διορισμό του Γενικού της Γραμματέα με λεπτομέρειες και σε πολλές ε, περιπτώσεις. Αυτές ήταν οι απαντήσεις ε, στα ερωτηματολόγια της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε σχέση με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε τον Απρίλιο και ως απάντηση των γραπτών ερωτήσεων του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, να πω καταρχάς ότι όλες οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται ε, αναρτημένες στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση των πολιτών. Ο Επίτροπος κ. Σέντιγκερ ήταν ε, παρόν στις δύο ολομέλειες και Επίσης, το Μάρτιο συμμετείχε σε μια κρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο Επίτροπος και, ε, και στην Ολομέλεια αλλά και στην ε, Ακρόαση απάντησε με λεπτομέρειες σε όσες ερωτήσεις του έγιναν. Ε, ο Επίτροπος Έτιγκερ τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού το Μάρτιο, διοργάνωσε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη διαδικασία επιλογής υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυτή έγινε σε 25 Σεπτεμβρίου και ήταν προσκεκλημένοι εκπρόσωποι όλων των θεσμικών οργάνων. Συζητήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός και οι λεπτομέρειες που αφορούν τον διορισμό των αξιωματούχων, ε, και ε, το πώς θα ενισχυθεί ο εσωτερικός ε, κανονισμός, πώς θα θωρακιστεί έτσι ώστε να, είναι, να έχει περισσότερη διαφάνεια και να επιτυγχάνεται αριστεία. Η συνθήκη παρόλα αυτά προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα θα έχουν την συνδρομή μιας ανεξάρτητης υπηρεσίες καθώς και ότι κάθε θεσμικό όργανο θα έχει αυτονομία σε ό,τι αφορά την ε, διοικητική του οργάνωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση του προσωπικού, ο εσωτερικός ε, κανονισμός των εξωματών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει όλες τις επιλημέρειες, όπως ακούσαμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλή τραπέζη, επιβεβαιώθηκε πω υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, ότι ο εσωτερικός κανονισμός που ε, νοδεύεται από νομολογία παρέχει ένα κατάλληλο και ισχυρό πλαίσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αυτονομία των θεσμικών οργάνων και ε, να έχουν εκείνα τη δυνατότητα να διορίζουν ε, σε διάφορες θέσεις προσωπικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν και ακολουθούν τα διάφορα θεσμικά όργανα για την επιλογή και τον διορισμό ανώτατων αξιωματούχων ενδεχομένως ε, διαφέρουν. Αλλά όλα τα θεσμικά όργανα ακολουθούν ε, τους ίδιους στόχους, δηλαδή θέλουν την πρόσληψη και την πρόθεση ταλαντούχων ε, υπαλλήλων με άρτια προσόντα. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ε, για τα υψηλόβαθμα στελέχη της, πάντοτε αυτό γίνεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό όπως αυτός έχει ερμηνευθεί από την ομολογία, καθώς και ε, με όλες τις σχετικές ε, διτάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας. Η, κυρία Ράιλι είχε πραγματικά εξαιρετική η εξαιρετικό επιτελείο. Η συνεργασία μα ήταν πάντα πάρα πολύ καλή. Έλαβε όντω ένα μεγάλο όγκο εγγράφων. Και όπω είπε και ο επίτροπο Έτινγκερ στην γραπτή του δήλωση το Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το γεγονό ότι η έκθεση με τι συστάσει δεν αμφισβητεί ούτε την νομιμότητα τη διαδικασία, ούτε όπω είπε μόλι τώρα η κυρία Ράιλι, την επιλογή των υποψηφίων ή του υποψηφίου. Αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε την απάντησή μας στις συστάσεις της διαμεσολαβήτριας και απαντήσεις αυτές θα σταλούν εμπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστές της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τον κύριο Σάρβαμα για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ουράιλη για αυτή την έκθεσή σας και για την παρουσίαση των συστάσεών σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα και υιοθέτησε ένα ψήφισμα στο ίδιο μηκο κύματο φέτος το 18. Οπότε χαίρομαι που επιβεβαιώνεται τα όσα εμείς είχαμε πει. σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερο feedback από την Κομισιόν. Οπότε η ερώτησή μου προς την Κομισιόν είναι τι μπορούμε να περιμένουμε από εσά και πότε. Ο κ. Σέλμαιρ, ο ίδιος προφανώς δεν θα πρέπει να ε, εμπλακεί στη συνέχεια που θα δοθεί. Όμως η, η ίδια η Επιτροπή, η Επιτροπή ελπίζω ότι θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρές κατευθύνες γραμμέ για τον διορισμό των υψηλών αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σεβάρμα. Ευχαριστώ γιατί ήσασταν γρήγορος καταρχήν. Παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε κύριε Οράιλη. Θα χρειαστεί να αποσιάσω για λίγο στην Επιτροπή Μεταφορών, αλλά θα επανέλθω αμέσω. Σε κάθε περίπτωση έχω εδώ ανθρώπους που θα ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την εκθέση σας κύριε Οράιλη. Δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Πρώτον, συγκρισιμότητα ανάμεσα στα δικά σας συμπεράσματα και με τα, με τα δικά μας. Δηλαδή να συγκρίνουμε τα συμπεράσματα. Ποια είναι τα, ε, η προστιθέμενη αξία των δικών σας συμπερασμάτων εναντί της δικής μας ε, γνωμοδότησης. Δεύτερον, εσείς, και με εξέπληξε αυτό, εστιάσατε αποκλειστικά στο διορισμό του Γενικού Γραμματέα. Προφανώς είναι ένα γεγονός το οποίο ξεσήκωσε τα πλήθη στις Βρυξέλλες και αλλού. Όμως, εμένα με εξέπληξε το γεγονός ότι ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα με την ευκαιρία του οποίου αντιληφθήκαμε δεν υπήρχαν κανόνες ε, αυτός ο διορισμός ε, συνέπεσε με τον διορισμό και τον αποδιορισμό, να το πω έτσι, ενός ολόκληρου καταλόγου διευθυντών και γενικών διευθυντών. Δηλαδή έγινε μετακίνηση τεκτονικών πλακών που επηρέασαν τελικά την, τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα. Πιστεύω ότι και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώσαμε ότι οι διορισμοί και οι αποδιορισμοί. Σε συνδυασμό με τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα δημιουργούν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Thank you, Ayala. Now, uh, for the ECR... Για το ECR δεν βλέπω κανέναν είτε από τους ε, φιλελεύθερους από τον, την ΚΟΕ δεν είστε από την Επιτροπή Κοντ, θα σας, θα σας δοθεί ο λόγος αργότερα. Ο κ. Στάς. Είναι εδώ ο κ. Στάς. Ναι. Mr. Tarrant, okay, you Ο κ. Τάραντ αντικαθιστάτε τον κύριο... Ναι, ωραία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπα στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, όταν συζητήσαμε το ίδιο θέμα, ο Φρίντριχ Ντεργκρόσε, ο περιβόητος, είπε κάποια στιγμή «Αν έχεις τη δυνατότητα να κατακτήσεις μια περιοχή, κάντο γρήγορα και μετά οι δικηγόροι και οι ιστορικοί θα ανακαλύψουν πολλούς λόγους για τους οποίους είχες δικαίωμα να το κάνεις». Έτσι έγινε και με, την, το διοσμό Σελμαέρ. Είναι ε, μια επίδειξη ισχύω. Κάνουμε ό,τι θέλουμε και αργότερα εξηγούμε μέσω κανονισμών, μέσω υπηρεσιακού κανονισμού και και λοιπά, γιατί μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα πρέπει όμως να μάθουμε το μάθημά μας, να διδαχθούμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι οι ψηφοφόροι δεν δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση για μας. Και αν ποτέ γίνω επίτροπος, κάτι που θεωρητικά μπορεί να συμβεί σε μια δημοκρατία, θα εγγυηθώ στον κύριο Σελμάιρ ότι η καριέρα θα τελειώσει με τον ίδιο με τρόπο παρόμοιο με αυτό που τελείωσε η καριέρα των προκατόχων του. <clears throat> Ωραία. Ο κύριος Ντε καιρό είχαμε να σας δούμε. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαία Διαμεσολαβητρία και την ομάδα της για την ε, έκθεσή της και τη σύστασή τους που ευθυγραμμίζεται με τους δικούς μας προβληματισμούς. Ο κ. Σέλμαερ ήρθε μόλις χτες για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και είχε δύο επιχειρήματα. Ε, είπε, ξέρω ότι δεν με αφορά εμένα προσωπικά η σύσταση αυτή, αλλά θα ήθελα να με είχε προσκαλέσει η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ε, ε, θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Ο κ. Σέτιγκερ μετά είπε ότι ανεξαρτήτως του πώς το οργανώνεται, το βασικό κριτήριο για το Γενικό Γραμματέα είναι να έχει την εμπιστοσύνη του Προέδρου της Κομισιόν. Οπότε, όπως και να έχουν τα πράγματα, εξαρτάται από τον Πρόεδρο της Κομισιόν. Θα ήθελα και γι' αυτό να ακούσω την άποψή σας. Τρίτη παρατήρηση. αν ε, προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο πλαίσιο του διοργανικού, στο, στο διοργανικό πλαίσιο, όλα αυτά θα γίνουν σε και κλεισμένο το θυρών. Ε, Μήπω όμω, επειδή το θέμα αυτό ξεσήκωσε πάρα πολύ την κοινή γνώμη, θα έπρεπε να γίνει κάτι δημόσια. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν, να ρωτήσω και τον εαυτό μα. Και εμεί θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Dennis. Ευχαριστούμε, Ντένις. Ε, η Βιωζίνη Γοσιέρ από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ, Σεσιλιά, ευχαριστώ την ε, διαμεσολαβήτρια για την παρουσίαση, για την ε, δουλειά σε αυτόν τον ευαίσθητο Βάκελο για ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μου δεν έχει επιληθεί καθόλου. Διαβάσαμε τις συστάσεις σας σχετικά με τη διαδικασία του ορισμού και προφανώς θα μπορούσε και να βελτιωθεί γιατί την άλλαξαν για να βολέψουν το διορισμό του κυρίου Ζέλμαια. Οπότε το ερώτημα είναι θέλουμε να συνεχίσουμε με την ουδετερότητα των διορισμών υψηλών θέσεων το οποίο συνάδει και με το ρόλο που υποτίθεται ότι διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τις συνθήκες. Ή θα πρέπει να υπαχθούμε σε μια καθαρά πολιτική προσέγγιση και διορισμό. Για οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ του προτύπου που υποτίθεται ότι ίσχυσε μέχρι τώρα και ενός προτύπου που θα έχει καθαρά πολιτικές αιτιάσεις και επιλογές, τουλάχιστον ας το πούμε. Γιατί αυτό υποσκάπτει τον θεσμικό ρόλο τη Κομισιόν. Εγώ υπήρξα δημόσια υπάλληλο, δημόσια λειτουργό πολλά χρόνια. Και πολλοί στεναχωριέ που μα λένε οι εκπρόσωποι τη Κομισιόν ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ότι υπάρχουν δημόσια διαθέσιμε απαντήσει και άλλα τέτοια. Υποσκάπτεται αυτή η ουδετερότητα επιλογών. Είναι θεμελιώδε ερώτημα του ρόλου που διαδραματίζει η Κομισιόν ω θεματοφύλακα των συνθηκών εδώ των συνθηκών και των κανόνων. Επίσης μας είπατε, μας αναφέρετε τέσσερις περιπτώσεις ε, κακοδιαχείρισης. Η Κομισιόν μας λέει ότι σεβάστηκε απόλυτα την νομιμότητα. Αλλά για τους πολίτες η καλή διαχείριση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Θα είχα πολύ μεγάλη περιέργεια γιατί θα είχε ποτέ το δικαστήριο να πει αν κάποιος προσέφευγε σε αυτό. Ε, Heidi για τους πράσινους. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη διαμεσολαβήτρια για μια πολύ σημαντική δουλειά που βοηθάει τους θεσμούς να πλησιάσουν λίγο τους πολίτες και ίσως ένα από τα διδάγματα που έχουμε από την υπόθεση αυτή, από την έρευνα αυτή είναι ότι πρέπει να έχουμε διαφανείς διαδικασίες διορισμού των ανώτατων αξιωματούχων. Και έχουμε και το έγγραφο που ετέθη στην Επιτροπή Γιούρι. Έχουμε το 99, με συγχωρείτε, 2, που δίνει ευρύτατες εξαιρέσεις για την διαδικασία του διαγωνισμού. Η δική μας ομάδα θεωρεί ότι οι γενικοί γραμματείς και στο Κοινοβούλιο και ίσως και οι γενικοί διευθυντές θα έπρεπε να μπορούν να διορίζονται μέσω μιας διαφανούς πολιτικής διαδικασίας. Κάτω από αυτή τη θέση όμως θα απαιτούσαμε μια απολύτως αντικειμενική διαδικασία και πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή το Προεδρείο συζητάει του διορισμούς εννέα διευθυντών. Και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην αντικειμενικότητα και διαφάνεια αυτών των διαδικασιών. Και αναφέρομαι στη σύστασή σα ότι δεν πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν ανταλλάγματα, παζάρι μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ πολιτικών κομμάτων ή ομάδων. Πώς θα φτάσουμε τελικώς όμως σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα έχουμε τέτοια. Αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά της Επιτροπής Πέτη, Πέτερ Γιάρ. Παρακαλώ, Έλικ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Διαμεσολαβήτριας. Συνοψίζοντας μπορώ να πω ότι η διαδικασία όχι δεν ήταν ιδανική. Μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Ναι, στην έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προσπάθ... έγινε προσπάθεια να εκτεθούν αντικειμενικά τα επιχειρήματα. Ε, και έχω μία ερώτηση παρόμοια με εκείνη που έκαναν οι συνάδελφοι. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Διότι έχουμε κοινή ευθύνη για αυτό που συνέβη. Και αυτό που συνέβη μάλιστα εξόργησε την κοινή γνώμη. Ε, και, και κλώνησε κάπως τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν φτάσει αναφορές πάρα πολλές οι οποίες ασκούν κριτική ακριβώς σε αυτό το ε, θέμα. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτές, ε, αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών και από την άλλη ε, υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας και κύρους ε, των θεσμών στις Βρυξέλλες. Τα θεσμικά όργανα οφείλουν να είναι αντικειμενικά και να χαρακτηρίζονται από ακαιρεότητα. Γι' αυτό λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε στο μέλλον να μην ξανάρθουμε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά. Ευχαριστώ πολύ Πέτερ έχει το Ευχαριστούμε πάρα πολύ στην την κυρία Οράιλη για αυτή την έκθεση και για την πολύ καλή συνεργασία. Συνεισφέρεται πολύ στη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Brexit. Η περίπτωση Μάρτι Σελμάιρ είναι πολύ κρίσιμη. Σηματοδοτεί το ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο από τους ε, πολίτες μας και να τους μην ε, ρίξουμε τους πολίτες μας τις αγκαλιές των λαϊκιστών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που όλα όσα προτείνει η διαμεσολαβήτρια. Αν η Κομισιόν δεν πάρει στα σοβαρά αυτές τις συστάσεις, θα διευκολύνουμε το έργο των εθνικιστών, που ακριβώς προσπαθούν να εντοπίσουν τέτοιου είδους ρογμές στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν να η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί με βάση τον εποτισμό. Έτσι κι αλλιώς η ίδια η διαμεσολαβήτρια συμπέρανε ότι ε, προσευλήθησαν οι διοικητικοί κανόνες ε, που ήδη είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν αντί να παίρνει αμυντική στάση θα πρέπει να αναλάβει δράση και να διορθώσει την κατάσταση. Χρειάζεται να διαθέτει μια διαφανή διαδικασία που δεν θα δημιουργεί υποψίες. Ελάχιστες εγγύησεις είναι το απολύτως απαραίτητο για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στις, στα θεσμικά όργανα. Κύριε Ράιλι, ποιο είναι ο πιο καλός τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα χωρίς να δώσουμε πυρομαχικά στους ευρωσκεπτικιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. On behalf of the Greens. Εκ μέρους των Πρασίνων, η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Ε, ο Σελμάιερ, από όσο ξέρω, μπορεί να μείνει σε αυτή τη θέση μέχρι να πεθάνει, μέχρι να πέσει από την καρέκλα του νεκρός. Αναφέρθηκε κάτι για την εμπιστοσύνη, για θέματα εμπιστοσύνης. Ναι, αν ήταν δικός μου βοηθός θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά αυτό που είπατε κύριε Ντεγιόγκ, να σας πω ότι πριν έρθω εδώ ήμουν 23 χρόνια βουλευτής στη Δανία και παρατήρησε ότι όλοι οι διορισμοί ήταν πολιτικοί διορισμοί στο κοινοβούλιο της, ε, ε, εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό δεν συμβαίνει στη Δανία. Αλλά εδώ θεωρείται δεδομένο ότι να ας πούμε αυτή η θέση θα πάει σε αυτή την πολιτική ομάδα, σε αυτή την επιτροπή θα βάλουμε ε, άτομα από εκείνη την πολιτική ομάδα. Δεν ξέρω αυτό για ποιους λόγους γίνεται, αλλά πραγματικά εξεπλάγει με αυτά που είδα. Και ορισμένοι Βρετανοί συνάδελφοι επίσης, τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Όλο το σύστημα εδώ ε, σοκάρει. Βέβαια η περίπτωση Σελμάρ είναι ακόμα χειρότερη, όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να κατανοήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι η θέση τους είναι να υπηρετούν ε, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χρηστή διακυβέρνηση σημαίνει ε, πως δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε στον πάτο πραγματικά. Στη Δανία υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο με ξέπλυμα χρήματος και εκεί ε, οι αρχές ανακάλυψαν ότι οι ρίζες πήγαιναν τόσο βαθιά που δεν μπορούσαν καν να κατανοήσουν ε, τι είχε συμβεί. Νομίζω πως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, κυρία Βαλένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη διαθεσιμότητα της διαμεσολαβήτριας ε, της ίδιας και όλης της ομάδας της να μας δίνει διαφημίσεις και εξηγήσει σχετικά με την ε, έρευνα αυτή. Νομίζω ότι η περίπτωση αυτή είναι μια απόδειξη του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρά κενά ελλείψεις αξιοπιστίας προς πολίτες και δεν μπορούμε να εκκλεισόμεθα με τις τάσεις κοινή γνώμης. Υπάρχουν πολλές αιτίε. Αλλά η περίπτωση του διορισμού του Γενικού Γραμματέα του Γιούνκερ, λέει η ομιλήτρια, αν το συνδυάσουμε με παρελθούς περιπτώσεις υπό τον Παρόσο των κυλιωμένων θυρών κτλ. Όλο αυτό το πράγμα επιβαρύνεται διαρκώς και η νομοποίησή του και η αξιοπιστία του βραχύνεται εξίσου διαρκώς. Υπάρχει ένα κώδικας διοντολογία ο οποίος δεν ακολουθείται. Υπάρχει κανονισμοί που δεν ακολουθούνται. Υπάρχει τακτική ενημέρωση που θα ήταν δημοκρατική οφειλή προ το κοινοβούλιο που δεν γίνεται. Εγώ δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας και να σας ε, ζητήσω να απαιτείτε διαρκώς τους απαραίτητους πόρους που χρειάζεται το, το οργανισμό σας ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί τόσο καλά. Ευχαριστούμε Άγχελα. Η κυρία Ήβη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την ε, διαμεσολαβήτρια O'Reilly για την εξαιρετική αυτή δουλειά, ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτήν συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοι να αντιμετωπίζουμε πολλά πολυάριθμα προβλήματα σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε εδώ. Αναφέρθηκε και η κυρία Βαλίνα στον κύριο Βαρόσο, τις περιπτώσεις του Ντράγκη, της ΕΚΤ, που συνεχίζει να είναι μέλος ιδιωτικών ομάδων όπως εκείνη των 30 κτλ. Και τώρα συζητούμε για το διορισμό του Ζελ Μάια, που όπως μας λέει ξεκάθαρα η δημοσιολαβήτρια μας, μας δίνει διάφορα παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων κακοδιαχείρισης όπως είπε και η ίδια στην επιλογή του ανθρώπου αυτού για γενικό γραμματεία δηλαδή στην ουσία διαμορφώνουμε τους κανόνες για να μας καλύπτουν και να μας βολεύουν ε, κατά το δοκούν αυτό είναι ε, επιβλαβές, ε, επιζήμιο για την αξιοπιστία της Κομισιόν και όλων των θεσμών με τρόπο πολύ ευρύτερο από αυτόν που γίνεται αντιληπτός. Εγώ λυπάμαι, αλλά τα λόγια που άκουσα από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σήμερα είναι απογοητευτικά και απλώς ε, σκοπεύουν να αποφύγουν την ερώτηση και να θολώσουν τα νερά. Σύμφωνα λοιπόν με την διαμεσολαβήτρια, ποιε είναι οι δράσεις που πρέπει να λάβουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πιο υψηλά πρότυπα ηθικά μεταξύ άλλων για τους υψηλούς θόκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η Πρόεδρο, για τη, συμμετοχή, για τη συμμετοχή σας στην συζήτηση αυτή. Βλέπω τώρα κάποια μέλη που δεν είχαν εγγραφεί στον κατάλογο. Αν κάποιος από εσά θέλει τώρα το λόγο. Θα σας δώσω από ένα λεπτό, αλλά παρακαλώ μην επαναλάβετε όσα είπαν οι προηγούμενοι. Προσπαθήστε για κάτι καινούριο ίσως. Ο κύριος Πυρίνσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω και εγώ μια ερώτηση για την κυρία Ράιλι. Μιλήσατε για συστάσεις και για την ανάγκη μιας ε, νέας ειδική διαδικασίας για ε, τέτοιους διορισμούς. Δεν θεωρείτε πως θα έπρεπε να γίνει και άλλη μια σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει δηλαδή τη δεύτερη σημασία στην ε, κοινή γνώμη. Διότι μου φαίνεται πως έχουν την ε, πεποίθηση πως είναι απολύτως, ε, πως κινούνται απολύτως στο πλαίσιο του νόμου με ένα μικρό ερωτηματικό ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ε, καλά το τι συνέβη, μάλλον έχει παρεξηγήσει κάποια πράγματα και ίσως ε, δεν έδειξαν τη δέουσα προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Κύριε Σαλαφράγκα, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε, ε, από τις λίγες φορές που έρχεστε στην Επιτροπή, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διακρίνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, το επίπεδο της πολιτικής ευθύνης, στο οποίο αναφέρθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι προφανές ότι η Κομισιόν ε, έχει ευθύνε απέναντι στην Επιτροπή μας. Δεύτερον, το επίπεδο της διαμεσολαβήτριας, η οποία ζητά η Κομισιόν να διαθέτει μια συγκεκριμένη διαδικασία για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα και πολύ καλό αυτό. Και τρίτον, η νομική ευθύνη. Μετά από την ομοδότηση της νομικής υπηρεσίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι ανεξαρτήτως του ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία. Νομικά στέκει, θέλω να πω, δεν έγινε παράβαση της νομοθεσίας. Νομίζω ότι το δίδαγμα είναι σαφές. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στους διορισμούς των υψηλών αξιωματούχων και των γενικών γραμματέων, αλλά όλα τα θεσμικά όργανα, πριν αρχίσουμε να προσπαθούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Γιατί και μέσα στο δικό μας το σπίτι έχουν γίνει παρατυπίες στους διορισμούς. Ο κανονισμός μας προβλέπει πολλές εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά το γενικό κανόνα Τη δημοσίευση μιας θέση που είναι ανακαλυφθεί. καλυφθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν γίνει τέτοιου είδους διορισμοί επανειλημμένω. και χαίρομαι που τουλάχιστον δεν αμφισβητούνται οι ικανότητε και τα προσόντα του Γενικού Γραμματέα της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Το δικό μου σχόλιο είναι ε, εκτό ότι έχουμε δυσκολίες με το πολιτικό σκηνικό γενικά στην Ευρώπη, έχουμε και άλλε πρόσθετε δυσκολίες. που συχνά ρίχνουν, ένα, ρίχνουν σκιές στην εικόνα μας. Κύριε Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διαφωνήσω με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα αποτελέσματα της ε, διοργανικής ανταλλαγής απόψεων. Και να σας θυμίσω ότι σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων κατέστη σαφές ότι ο ειδικό ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαινόταν στην επιλογή ε, του προσωπικού της. Ε, δεν έγινε, όπως σας είπα, ε, προκήρυξη, δεν έγινε ανοιχτός διαγωνισμός για το Γενικό Γραμματέα, αλλά και για πολλούς διευθυντές. Οι θέσεις αυτές καλύφθηκαν με εσωτερικές ε, μεταθέσεις. Το καταστατικό όμως ε, και ε, προβλέπει αυτές τις εξαιρέσεις καθώς και η νομολογία τονίζει αυτές τις εξαιρέσεις. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία καταξαίρεση η οποία ισχύει και ακολουθήθηκε. Δεν θέλω τώρα να ανακατέψω πράγματα του παρελθόντος, αλλά αυτές οι απαντήσεις που μας δώσατε δεν ισχύουν. Μας είπατε ότι μας ενημερώσατε, εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση. Ε, και σε ό,τι αφορά το έργο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, πρέπει να, πρέπει να το αποδεχτείτε και εσείς ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και δεν μπορείτε να το αρνείστε. Εσάι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάβαλ, θα ήθελες το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Ράιλι για την παρουσίασή της, διότι για μένα κατέστη σαφές ότι ο εσωτερικός κανονισμός έχει κάποιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά τον ε, διορισμό υψηλοβαθμών αξιωματούχων. Μας λείπει ένα πλαίσιο και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τα θεσμικά όργανα, ε, το οποίο πλαίσιο θα επιτρέψει την ε, εφαρμογή των κανονισμών σε ό,τι αφορά τους ε, διορισμούς αυτούς. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Απρίλιο του 2018 είναι ξεκάθαρο. Ω θεσμικό όργανο πρέπει να έχουμε την εντολή για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και να προ βλέπουμε σε μια ε, βελτίωση της ε, διοργανικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, κάλυψη τέτοιων θέσεων. Ευχαριστώ. Χρειάζεται όντως να διασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί του προσωπικού και το καταστατικό θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Είναι κοινή λογική. Υπάρχουν κανονισμοί, αλλά η λογική είναι αυτό που λείπει. Ας ελπίσουμε λοιπόν πως θα πριτανεύσει η λογική ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη φορά που θα προκύψει κάτι τέτοιο. Και ελπίζω να μην χρειαστεί καν δηλαδή να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια που ήρθε. Και φυσικά, φυσικά θα σας δώσω το λόγο έτσι ώστε να ε, αντιδράσετε σε όλα αυτά που ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Να ευχαριστήσω ξανά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεργασία που έδειξε σε αυτήν την ε, αδιάκοπη ανταλλαγή γράφων που έλαβε χώρα το καλοκαίρι ε, σε ό,τι αφορά τα προσόντα του κυρίου Σελμαέρη να πω ότι δεν αμφισβήτησα την νομιμότητα του διορισμού του. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το δικαστήριο. Αυτό που ανέφερα ήταν ορισμένες ε, παράμετροι ε, που αφορούν την νομιμότητα, οι οποίες παράμετροι ίσως ε, να τραβήθηκαν λίγο στα άκρα. Η έρευνα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατέληξε σε πορίσματα και συστάσεις τα οποία λίγο πολύ συμφωνούν με αυτά που ακούσαμε λάβαμε μεγάλο όγκο εγγράφων και οι έρευνές μας είναι βασισμένες σε στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες μετά να τα ε, διαβάσουν και να εξάγουν μόνοι του συμπεράσματα. Από όσο γνωρίζω από το επιτελείο του κυρίου Σελμάιερ, απάντησε σε ερωτήσεις που του έγιναν αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έγινε μια παρεξήγηση. Υπήρχε η εντύπωση ότι ε, ερευνούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τον ίδιο τον ε, κύριο ε, Σελμάιρ. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έλαβε μεγάλε διαστάσει και πολλή δημοσιότητα, περισσότερη από ότι αν ήταν κάποιος άλλος και όχι ο κύριο Σελμάιρ, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ε, εστάλησαν αρκετέ εκατοντάδε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και ο κύριος Σέλμαιρ έδωσε απαντήσεις οι οποίες εστάλησαν σε εμάς και πάνω σε αυτές ε, εργαστήκαμε. Κύριε Ντεγιόγκ, συμφωνώ μαζί σας. Δεν μπορείς να διορίζεις έναν ανώτατο αξιωματούχο χρησιμοποιώντας αλγόριθμο. Πρέπει να υπάρχει ε, και κάποια συμβατότητα, πρέπει να υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας όταν επιλέγεις. Όμως, αυτό ίσως ίσως ταιριάζει περισσότερο για θέσεις ε, του, στο επιτελείο ενός επιτρόπου παρά για τον Γενικό Γραμματέα της ίδιας της Επιτροπής. Προσπάθησα να δω πώς έγινε αυτός ο διαχωρισμός από, την, ε, από τη θέση του επικεφαλής του επιτελείου, από τη μία που είναι, πολύ, είναι άκρος πολιτική ε, και από την άλλη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα που δεν είναι. Νομίζω πως ο διορισμός αυτός είχε το εξής πρόβλημα. Για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα χρησιμοποίησαν ε, μέσα τα οποία βοήθησαν τον κύριο Σελμάιερ να καταλάβει αυτή τη θέση. Και αν δεν κάνω λάθος, η θέση αυτή είχε μείνει άδεια για κάποιους μήνες. Τώρα, σε τη φορά τις ερωτήσεις που έγιναν για τις συστάσεις μου, να σας πω ότι πράγματι έκανα συγκεκριμένες συστάσεις για το διορισμό ε, του Γενικού Γραμματέα, για τη θέση αυτή και όταν ερωτήθηκα εάν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συστάσεις σε ευρύτερο πλαίσιο, να πω ότι είμαι κάπως διστακτική για κάτι τέτοιο. Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες για τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Κομισιόν, Μίλησα σε μια επιτροπή, στην Επιτροπή Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν δεν κάνω λάθο. Και ε, παρά το γεγονό ότι αυτά που υπαφορούσαν το Γενικό Γραμματέα τη Κομισιόν, ε, ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε ευρύτερα. Φυσικά δεν είμαι εγώ αυτή που θα κάνει υποδείξεις για το πώς ε, θα ε, είναι ο γενικό ο ιστορικός κανονισμός, πώς θα γίνονται αυτά. Μπορώ να κάνω συστάσεις όμως. Και έγινε και μια άλλη ερώτηση. Νομίζω ο κύριος Πυρίνσκι έκανε την ερώτηση αυτή για τις συστάσεις ε, ε, του να λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κοινή γνώμη από εδώ και στο εξή. Μια από τις ερωτήσεις που έκανα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν και αυτή. Αρχικά, ήθελα να να δω τις αντιδράσεις, να δω τις αντιδράσεις του κοινού και να δώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρόνο για να επεξεργαστεί όλες αυτές τις πληροφορίες. Ε, πολλά ερωτήματα ήταν αναπάντητα, αλλά ήθελα να τους δώσω χρόνο να αναλογιστούν ε, αυτές τις ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν το έκαναν και αυτό είναι κρίμα. Νομίζω έγινε ένα σχόλιο ότι είχε ανέβει και μια δημοσκόπηση από το Ευρωβαρόμετρο λίγο μετά το διορισμό Σελμάιερ και έδειξε ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι φυσικά καλό. Αλλά και ότι ο διορισμός Σελμάιερ δεν είχε κάτι το αμφιλεγόμενο. Όμως αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τη χώρα ε, που γίνεται μια τέτοια δημοσκόπηση. Στη Βρετανία, ας πούμε, υπήρχαν άλλες απόψεις. Όλα αυτά, αργά ή γρήγορα, φτάνουν στα μέσα ενημέρωσης. Και το γεγονός είναι ότι τα θεσμικά όργανα, εφόσον προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις, πρέπει να ε, τις αντιμετωπίσουν. Φυσικά, να σας πω ότι θαυμάζω το επίπεδο δίκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ υψηλό και φυσικά αυτό εξυπακούεται λόγω του ρόλου τους, του θεσμικού τους ρόλου. Αλλά όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να λειτουργούν υποδειγματικά. Μετά μου έγιναν συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Όπως σας είπα, ε, διστάζω να ε, τοποθετηθώ και να γίνω απόλυτη, ούτε θέλω να κάνω υποδείξεις, αλλά νομίζω πως λίγο πολύ όλα αυτά που είπα μπορούν να καλύψουν αυτήν την ερώτηση. Σας ευχαριστούμε για την ε, ετοιμότητά σας να έρθετε εδώ, να μας ε, εξηγήσετε τα πορίσματα και τα συμπεράσματά σας και να συνομιλήσετε με εκπροσώπους τριών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω τους συμπροέδρους, Παύελ Ινιεμπόρε, και όλους εσάς. Διακόπτω την συνεδρίαση για δύο λεπτά για να μπορέσουμε να αναδιοργανωθούμε.